δύσκολο να βρεθεί η βέλτιστη λύση μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων. Ελπίζω να καταφέρουμε να τη βρούμε πέρα τη συζήτηση και αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κοινή συζήτηση Σέγγεν. Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν και προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Πρώτα θα μιλήσουν οι εισηγητές. Καταρχάς ο κύριος Κάρλος Κοέλιο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές φτάσαμε σε ένα συντονισμό, σε μια συμφωνία για το πακέτο Σέγγεν. Ε, δεν είναι απόλυτη ε, τα όσα εμείς είχαμε ζητήσει, γιατί μας αρνήθηκαν την νόμιμη και θεμητή συναπόφαση, αλλά πρόκειται για σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα κανόνε και την διαχείριση του συστήματος Σέγγεν. Προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθερα. Επιτρέψατε μου να υπογραμμίσω τα εξή. Καταρχήν, επιλέξαμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ο μηχανισμό αξιολόγηση ε, δεν θα είναι πλέον ε, διακυβερνητικό, αλλά θα είναι ευρωπαϊκή φύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίζει ρόλο απλού παρατηρητή και για τον γενικό συντονισμό επίση θα τον αναλάβει εκείνη και για την παρακολούθηση τη λειτουργία του σήματο. Θα είναι υπεύθυνη για τη λήψη των περισσότερων αποφάσεων σε σχέση με το ετήσιο και πολιτέ πρόγραμμα για την προετοιμασία ε, επιτόπου επισκέψεων και για τις συστάσεις. θα προτείνει επίση συστάσει για διορθωτικέ δράσει που θα εγκριθούνται στη συνέχεια από το Συμβούλιο. Έπειτα θα συμπλέκονται διάφορε υπηρεσίε και θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν αγνοούμε τα εσωτερικά σύνορα. Προβλέπεται η δυνατότητα να εκτιμάται αν θα γίνονται ή όχι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Σε συγκεκριμένε περιπτώσει, όπω αυτέ που αντιμετωπίσαμε τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη που κάποιε φορέ εμπνεύστηκαν από από εθνικές ατζέντε ε, και που επιβλήθηκαν από κόμματα ακράς δεξιάς. Έπειτα καταργήσαμε τα διπλά μέτρα και σταθμά που ισχύουν σήμερα. Από τώρα και στο εξή, οι χώρε υποψήφιε και οι χώρε που είναι ήδη μέλη του ΣΕΝΚΙ θα πρέπει να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με ε, του ίδιου κανόνε. Οι αρχέ του ΣΕΝΚΙ θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ αυστηρά, όχι μόνο πριν αλλά και μετά την ένταξη. Η έλλειψη αυστηρότητας του ισχύοντος ε, μηχανισμού θεωρηθεί, οδήγησε στο να ε, υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα όσον αφορά την αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση δίνει δυνατότητα να γίνονται έλεγχοι επιτόπου στα εσωτερικά σύνορα χωρίς προειδοποίηση και μάλιστα και στα εξωτερικά σύνορα. Έτσι δίνουμε μεγαλύτερη βάση στο σύστημα αξιολόγησης. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Υπάρχει μια αξιολόγηση μεταξύ ίσων, ενώ το σύστημα ε, επαλήθευσης και αξιολόγησης θα επιτρέπει πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση. Θα συμπληρώνονται έτσι οι άλλοι κανόνες του Σέγγιν και έτσι θα γίνεται διορθωτική δράση έτσι ώστε να προβλεφθεί και να διαλυθεί αυτό το αίσθημα της ατιμορρησίας. Έπειτα, ενισχύσαμε τον δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγγυηθήκαμε την πρόσβαση στα έγγραφα. Θα ενημερώνεται διαρκώ το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τη διαδικασία και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα για το Frontex, για το πολυμερέ και ετήσιο πρόγραμμα ε, αξιολόγηση ε, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ε, ελλείψεις. Ε, θα μπορεί να δει επίσης τις απαντήσεις των ε, κρατών μελών στις, ε, στα ερωτηματολόγια. Πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια που, γιατί προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε πρόσβαση σε κανένα έγγραφο σε σχέση με το Σέγγεν. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγαλύτερο έλεγχο για τις μελλοντικέ πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα. Υπάρχει έτσι λοιπόν καλύτερο συντονισμός και μέσα στο πλαίσιο του εγγράφου. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλσορμα, αλλά και την ε, Ιρλανδική Προεδρία για τη συνεργασία τους. Αυτή η συμβιβαστική έχει, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού αξιολόγησης ε, με μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότητα. Ε, ε, ζητώ λοιπόν την υποστήριξή σας για αυτή τη συμβαστική λύση και οφείλεται στην σταθερή και έντονη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές που ποτέ δεν αρνήθηκαν τη στήριξή τους ακόμα και αν προέρχονταν από διαφορετικές, ε, από διαφορετικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ. Τέσσερα λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε χρόνο γίνεται μία έρευνα για το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 50% λένε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη μετακίνηση και έχουν κάθε λόγο να το ισχυρίζονται αυτό. Στην Ευρώπη όπου για δεκαετίες οι άνθρωποι, οι οικογένειες ήταν χωρισμένοι από σύνορα βρίσκονται πλέον σε μία περιοχή όπου είναι ελεύθερη μετακίνηση και έτσι αισθάνονται ότι ζουν σε ένα μεγάλο σπίτι. Επίση, είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσουν τα οικονομικά ωφέλη που απορρέουν από τι επιχειρήσει μα. Γιατί λοιπόν χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνο για να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο τόσο πολύ επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Η απάντηση είναι απλή αλλά και περίπλοκη παράλληλα. Υπάρχουν ε, λαϊκίστικες απόψει σε πολλά κράτη-μέλη, γίνονται εκλογέ σε διάφορα κράτη-μέλη και αυτό επηρέασε την συμπεριφορά ορισμένων κυβερνήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει να που καταλήξαμε. Μιλάμε για τον ε, κώδικα του Σέγγεν που πλέον ε, καθορίζει σαφείς ε, στόχους για ε, συγκεκριμένες καταστάσεις ε, για τον ε, επανέλεγχο στα σύνορα, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις. Ομολογώ λοιπόν ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να υπάρχουν αποφάσεις για την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η εποχή. Πρέπει να πούμε ότι κατορθώσαμε να εισάγουμε την κοινοτική διάσταση, επιπρόσθετες εγγύησεις, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση των μηχανισμών. Οι δυνατότητες που υπάρχουν τώρα να επανέλθουν ε, ε, οι έλεγχοι στα σύνορα διευκρινίστηκαν και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ε, τεστ της αναλογικότητας για να μετρώνται οι επιπτώσεις, να γίνονται διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, κυρίως σε αυτά που επηρεάζονται από την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων, να λαμβάνονται υπόψη οι γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε ζητηθεί, υπήρξε το αίτημα του Συμβουλίου να επανέλθουν οι έλεγχοι. Αυτό το αίτημα εκφράστηκε προ την Κομισιόν πριν από δύο χρόνια. Αυτό όμω θα είναι μόνο η έσχατη λύση ε, σε ειδικέ καταστάσει ε, όταν διαπιστωθούν ότι υπάρχουν πραγματικά κενά στου ε, συνοριακού ελέγχου. Στην περίπτωση όμω αυτή η πρόταση θα έρθει από την Επιτροπή μετά από εντελεχή αξιολόγηση. Υπάρχουν λοιπόν έλεγχοι που θα πρέπει να φέρουμε τα Επανήλθε ένα συγκεκριμένο εδάφιο, μια αιτιολογική σκέψη για να διατηρηθούν οι υποχρεώσει του 2011. Ε, Πολλέ, ε, πολλοί πήκοοι τρίτων χωρών δεν πρέπει αυτομάτως να θεωρούνται απειλή στην ε, εσωτερική ασφάλεια. Η συνολική περίοδος κατά την οποία μπορούν να επανεισαχθούν οι συνοριακοί έλεγχοι με βάση την απειλή στην εσωτερική ασφάλεια, αυτή η χρονική περίοδος δεν μπορεί να ξεπερνάει του τους δύο μήνες. Η Κομισιόν οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον μία ετήσια έκθεση για την λειτουργία μιας περιοχής χωρίς εσωτερικούς ελέγχους. Και αυτή η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την επανεισαγωγή των εσωτερικών ελέγχων ε, κατά μία συγκεκριμένη χρονιά. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια και για την έκθεση του κυρίου Κοέλιο, όπου είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Εδώ το πραγματικό επίτευγμα είναι ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο μηχανισμός βασίζεται σε έκθεση ομοτήμων. Η Επιτροπή στο μέλλον θα είναι αρμόδια για όλες τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται είτε με τη μορφή της Επιτροπολογίας είτε θα τις λαμβάνει και μόνη της. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει ε, προτάσεις ε, μετά από συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι υιοθετήθηκε μια κοινή πρόταση από τους τρεις θεσμούς και οποιαδήποτε πρόθεση της Κομισιόν που θα αξιολογεί το μηχανισμό πρέπει να κατατίθεται στο Κοινοβούλιο για διαβουλεύσεις. Αν εγκριθεί αυτό, τότε αυτομάτως θα υπάρχει προηγούμενο γιατί ε, πρέπει το ε, άρθρο 70 να λαμβάνεται υπόψη που είναι η υποχρέωση και η δέσμευση προς ε, διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Συμβουλίου η κυρία Κράιτον. Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, εξ ονόματος της Ιρλανδικής Προεδρίας θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που καταφέραμε να καταλήξουμε στη συμφωνία για το νομοθετικό ε, πακέτο για την διακυβέρνηση στη Σέγγεν το Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο του 2011 στα συμπεράσματά του να βελτιωθεί η διαδικασία της Σέγγεν και να μπορεί να ανταποκρίνεται και σε έκτακτες συνθήκες, κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να θέσει κινδύνο το όλο σύστημα Σέγγεν. Αποφασίστηκε βέβαια να προστατεύσουμε την ε, διαδικασία της ελευθερίας της μετακίνησης και προσπαθήσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα την ελεύθερη μετακίνηση. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτέγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της τελευταίας δεκαετίας. Η ελευθερία κυκλοφορίας ε, ε, είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινή πραγματικότητα για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και τους υπηκόους των τρίτων χωρών που βρίσκονται στον ευρωπαϊκό χώρο ως επισκέπτες οι μόνιμοι κάτοικοι. Γίνονται χιλιάδες ταξίδια, εκατομμύρια ταξίδια κάθε χρόνο και ε, η δυνατότητα αυτή είναι ένα από τα πιο σημαντικά ωφέλη σύμφωνα με τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν καταφέραμε να ενισχύσουμε τις διαδικασίες για να έχουμε καλύτερη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης ε, Σέγγεν μαζί με τον κατάλληλο μηχανισμό ανταπόκρισης συγκεκριμένων απειλών θα συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το στόχο και ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη διαφάνεια των ε, διαδικασιών. Συνειδητοποιώ βεβαίως πλήρως ότι οι διαπραγματεύσει για τα μέτρα αυτά δεν ήταν εύκολες. Ξεκινήσαμε με τη ε, διάσταση απόψεων για τη νομική βάση για τη ε, διαδικασία της Σέγγεν, αλλά ε, πλέον αυτό αντιμετωπίστηκε και μάλιστα με επιτυχία. Χαίρομαι διότι καταφέραμε να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων προεδριών και να βρούμε μια σωστή άγουσα από κοινού. Έχουμε υπερκεράσει δυσκολίες και έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο το δυνατόν περισσότερο για, για τα δύο μέτρα. Η συνολική συμφωνία περιλαμβάνει και μια κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονό το οποίο καταστη... Ε, ε, ε, καθιστά σαφέ ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα υποβάλλεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συμβουλευτικού λόγου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η άποψή του πλήρω πριν την έγκριση ενό τελικού κειμένου, όπω συνέβη και με την παρούσα πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ειλικρινά εκ βάθους καρδίας για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί μας προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αναγνωρίζω ότι η πρόταση αξιολόγηση ε, ε, εγκρίθηκε χθε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμο για να εγκριθεί το πλήρε πακέτο αύριο στην Ολομέλεια. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω του εισηγητέ για τι δύο νομοθετικέ προτάσει, την κυρία Ρενάντε Βέμπερ και τον κύριο Κάρλιο Σκοέλιο, οι οποίοι με τη δέσμευσή τους και τη σκληρή τους εργασία κατάφεραν πραγματικά να διασφαλίσουν ε, τη συμφωνία. Η συνεισφορά σας λοιπόν εκτιμάται ιδιαίτερως από την Προεδρία μας και από το Συμβούλιο εν γέννη, όπως ε, ε, φυσικά γίνεται και με τα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ακούσω την ε, συνεισφορά των ε, περισσότερων ευρωβουλευτών. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη όμως. Δυστυχώς πρέπει να φύγω νωρίτερα. Υπάρχει τριμερής διάλογος για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επίτροπος Μάλστρομ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη, η ε, κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Βερβουλευτές. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο στην ίδια αίθουσα βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ε, υπήρχαν πολύ έντονα συναισθήματα και εντάσεις ανάμεσα στα, διάφορα, στα τρία θεσμικά όργανα. Σήμερα ένας χρόνος έχει περάσει και χάρη στις εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο που παίξατε πολύ ισχυρό και επικοδομητικό ρόλο και τις διάφορες προεδρίες, την Κυπριακή και την Ιρλανδική, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία για τη διακυβέρνηση του Σέγγεν. Έχουμε τώρα το μέσο που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε το Σέγγεν και γι' αυτό η Κομισιόν μπορεί πλήρως να στηρίξει τον συμβιβασμό που επετέφει. Θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές Κάρλος Κουέλιο και Ρενάτε Βέμπερ. Ξέρω πόσο σκληρά δουλέψατε. Μαζί με τους κοιόδες εισηγητές και τους συνεργάτες σας ήταν φανταστικοί σε όλη αυτή τη μακρά πορεία. Ο συμβιβασμός που πετέφθη, όπως είπατε, θα επιφέρει μεγάλες βελτιώσεις σε σύγκριση με το ίσχυον σύστημα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ήδη ένα ε, σύστημα για να χρησιμοποιήσουν το κεκτημένο του Σέγγεν τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφέ πω δεν πρόκειται για μηχανισμό που απολύτω χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα νέο που εξασφαλίζει ότι ο χώρο χωρί εσωτερικού συνοριακού ελέγχου προστατεύεται καλύτερα και είναι καλύτερα εξοπλισμένο για να εντοπιστούν οι ελλείψει σε πρώιμο στάδιο και να εξασφαλίσει τη λήψη καταλήλων μέτρων, καθώ και να δίνεται η κατάλληλη συνέχεια. Αυτό ο αναθεωρημένο μηχανισμό θα προσφέρει αυτό και θα έχει, περιλαμβάνει περισσότερη διαφάνεια. Η Κομισιόν έχει συντονιστικό ρόλο, η αξιολόγηση θα γίνεται από την Κομισιόν μαζί με τους εμπειρογνώμενου των κρατών μελών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ε, ανακύψουν σοβαρές ελλείψεις, ο προτινόμενο μηχανισμός προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπω για παράδειγμα την αναδίπλωση ε, ε, των ευρωπαϊκών συνοριοφυλάκων της Frontex. Επίση, προβλέπεται το σύστημα να ανταποκρίνεται σε περιστάσεις όπου, υπάρχουν συστάσεις, όπου δεν αρκούν μάλλον οι συστάσεις για άμεση δράση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι, μόνοι, οι διαρκείς και μόνιμε πιέσει σε ένα νέο σύστημα επιτρέπει συναπόφαση για την προσωρινή επανεισαγωγή εσωτερικών συνοριακών ελέγχων. Σταφώ δηλώνατε όμω ότι θα είναι ένα έκτακτο μέτρο ω τελευταίο καταφύγιο σε μια πραγματικά κρίσιμη κατάσταση και αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο ώστε να εξασφαλιστεί η επίλυση προβλημάτων ενώ θα ελεγχιστοποιηθεί ο αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία. Το νέο σύστημα Επίση, ε, δίνει πολλά πλονεκτήματα στο Κοινοβούλιο που θα έχει αυξημένε δυνατότητε επιρροή στη λειτουργία του χώρου Σέγγεν γιατί θα λαμβάνει όλε τι σχετικέ πληροφορίε και το Συμβούλιο και η Κομισιόν εξέφρασαν την πολιτική του βούληση να, να συμβουλεύονται το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν. Το η κοινή δήλωση που θα συνοδεύει την απόφαση δηλώνει σαφώ ότι οποιαδήποτε σύσταση τη Κομισιόν για τροποποίηση του συστήματο, θα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και ότι η γνωμοδότησή του θα λαμβάνεται υπόψη πλήρω όσο αυτό είναι δυνατόν, πριν την υιοθέτηση του τελικού κειμένου. Νομίζω πως με αυτή τη διευκρίνηση, αυτή την ενίσχυση των ε, μέσων που υπάρχουν θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη συμβιβαστική που πετύχαμε και όπως και στην προηγούμενη συζήτηση που πολλοί από σας παρακολουθήσατε δείχνει πως όταν πραγματικά ε, συντονιστούμε τα τρία θεσμικά όργανα ε, ωφελούν, λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα θα προχωρήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος είναι ο κύριος Βέμπερ για το ΕΛΚΑ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, η Ιρλανδική Προεδρία αυτή την εβδομάδα ολοκλήρωσε δύο σημαντικούς φακέλους στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, το άσυλο και τη Συμφωνία Σέγγεν. Κατόπιν του, του για μας η Ιρλανδική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και σας συγχαίρουμε. Και ελπίζουμε να τα καταφέρετε και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, να προχωρήσετε και εκεί με τα θέματα της χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό ακόμα θεωρεί το Σέγγεν ε, ένα πολύ σημαντικό χώρο. Η εισηγήτριά μα, η κυρία Βέμπερ, αλλά και ο κύριο Κοέλιο δούλεψαν πάρα πολύ καλά και του ε, συγχαίρουμε. Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί δημαγωγοί και στη Γαλλία και στην Ουγγαρία και στην Βουλγαρία που ε, επιθυμούν ως δημαγωγοί τη δεξιάς να πείσουν τους πολίτε ότι είναι περιττό το Σέγγεν. Εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε ανοιχτό το πεδίο. Το Σέγγεν φέρνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και αυτό θέλουμε να πετύχουμε με την τροποποίηση του δικαίου. Αυτοί λοιπόν οι λαϊκιστές επιθυμούν να επαναφέρουν την Ευρώπη σε ένα ζωφερό παρελθόν. Ε, πρόοδος υπάρχει και στην αξιολόγηση. Το είπαν αυτό οι συγητές μας. Και κυρία Επίτροπε θέλω να σας πω ότι χαίρομαι για τις εκθέσεις που θα υποβληθούν από ουδέτερους συντάκτες. Χαίρομαι που θα έχουμε ουδέτερες εκθέσεις όπου κάποιοι Υπουργοί Εσωτερικών δεν θα χαρούν και πάρα πολύ ότι θα πρέπει να υποβάλουν την αξιολόγησή τους ε, στην Frontex ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμως θα ενισχύσει το σύστημα. Αρνητικό είναι βέβαια το ότι τα δικαιώματα συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναγνωρίστηκαν στην αξιολόγηση. Και εξακολουθώ να μην καταβέλω γιατί μπλοκάρει το ε, Συμβούλιο. Το να επιθυμείτε να υπεραμεινθείτε πάση θυσία των δικαιωμάτων του Συμβουλίου, αυτό για μένα σημαίνει ότι δεν επιθυμείτε τη διαφάνεια και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον θα αγωνιστεί ε, αποφασισμένα για τα δικαιώματα των Ευρωβουλευτών και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, ο κύριος Ενσιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους δύο εισηγητές ε, για την ε, ε, επιμονή με την οποία εργάστηκαν για να φτάσουν στο σημερινό αποτέλεσμα. Και να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η συμφωνία ε, για ε, το κεκτημένο του ε, Σέγγεν απέχει κατά πολύ από αυτό που πρότεινε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως το πρώην μοντέλο που λειτουργήσε, το μοντέλο εκείνο κατ' ουσίαν περιόριζε την ελεύθερη μετακίνηση στο χώρο Σέγγεν. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι στο μέλλον δεν ε, ε, θα πρέπει να αποφεύγουμε τις καταχρήσεις. Τα σύνορα του χώρου Σέγγεν πολλές φορές αξιολογήθηκαν καταχρηστικά. Μέχρι σήμερα είχαμε δύο διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης. Ένα σύστημα που λειτουργούσε πάρα πολύ χαλάρα και ένα άλλο σύστημα για τις υποψήφιες χώρες. Αυτά λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά οδήγησαν σε ακραίες και παράδοξες καταστάσεις όπου χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία ε, μέχρι τώρα δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο χώρο του Σέγγεν παρότι ε, για τις ε, χώρες αυτές ισχύουν ιδιαίτερα αυστηροί κανονισμοί. Άρα δηλαδή παντού θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Όσον αφορά στην αξιολόγηση πρέπει να ισχύσουν ευρωπαϊκά κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και η Επιτροπή ε, θα συζητήσει και για την ε, επαναφορά ε, των ελέγχων στα σύνορα. Νομίζω λοιπόν ότι η Frontex πρέπει να έχει σαφέστερα καθήκοντα, αρμοδιότητες που δεν είχε μέχρι σήμερα. Εφ' θα υπάρχει ένα σχέδιο παρακολούθησης που θα το συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως όταν θα διαπιστώνεται ότι έχει παραβιαστεί το κεκτημένο Σέγγεν. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την ε, βραχία, την προσωρινή επαναφορά ελέγχων στα σύνορα, οποτεδήποτε διαπιστώνει κάποιες παραλήψεις. Επίσης ε, πιστεύω ότι η ε, πρόσβαση σε όλες τις ε, τράπεζες δεδομένων αυτό αποτελεί μια βελτίωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δική μου εν πάση περιπτώσει τη χώρα αλλά και για άλλες χώρες εκτός του χώρου Schengen όλα αυτά τα μέτρα κρίνονται ανεπαρκή εάν δεν εισαχθούν και κανόνες για την συμπερίληψη νέων ε, χωρών ε, στο χώρο του Σέγκεν. Επαναλαμβάνω, η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρεμποδίζεται εδώ και δύο χρόνια, παρότι αυτό αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Έχω λοιπόν μία παράκληση. Επιθυμώ να προτείνω στο Κοινοβούλιο ένα νέο μέτρο που να αφορά στην ε, συμπερίληψη νέων κρατών στο χώρο του Σέγγεν. Η συγγήτρια, η κυρία Βίμπα, έχει το λόγο. Νομίζω πως είναι λάθος ε, να ξαναμιλήσω, αλλά το υποφελούμε για να ευχαριστήσω πολύ την Ελλαδική Προεδρία, επειδή η ε, Υπουργό θα φύγει. Και πραγματικά και ειλικρινά σας ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλατε για να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση. hát äh, ε, θέλει να απαντήσει. Ωραία, από μακριά ευχαριστείτε, εντάξει. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μετά από αυτή την ε, σύντομη διακοπή κυρίας Ντάνοκα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργέ, αγαπητοί Επίτροπε, συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, Κοέλιο και Βέμπερ, τους εισηγητές μας, Κοέλιο και Βέμπερ, για τις ε, ε, πολλές τους προσπάθειες να διατηρηθούν οι θέσεις του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή πριν από ένα χρόνο. Είναι λυπηρό που αυτές οι προσπάθειες δεν ε, βελτίωσαν την επιτυχία. Στην αρχική προσπάθεια ε, προτάθηκε ένας μηχανισμός που θα βασίζεται στην Ένωση για την προσωρινή εισαγωγή ελέγχων και την αξιολόγηση του Σέγγεν. Επίσης, ήμασταν αντίθετοι αντίθετη στην αναθεώρηση της νομικής βάσης για την νομοθεσία Σέγγεν ε, που απέκλειε το Κοινοβούλιο από την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων ακόμα και αν η Κομισιόν απέφυ, ε, δεν κατάφερε να υποστηρίξει την προσέγγιση της Ένωσης η τελική απόφαση για μια εθελοντική συμβιβαστική δεν είναι η καλύτερη λύση και τέλος η αναφορά στην παράνομη μετανάστευση δεν είναι αποδεκτικά για μας αν λάβουμε υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε στις 29 Μαΐου ε, την συμφωνία της 29 Μαΐου. Αυτό το αποτέλεσμα σαφώς είναι ε, λυπηρό για την ακαιρεότητα του Σέγγεν. Ο κύριος Βαντάλεν, χωρίς μικρόφωνο. Let us try another one. Δοκιμάστε κάποιο άλλο μικρόφωνο. This is better. Yeah. Μ' ακούτε τώρα. Ωραία. Τα ξαναλέω. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία αυτή για την νομοθεσία Σέγγεν επιτρέπει να γίνονται έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αλλά λέει ταυτόχρονα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ιερή. Η έλεγχη αυτή θα είναι εξαίρεση, παραδείγματος χάρη αν υπάρχει τρομοκρατική απειλή. Κατ' εμέ αυτή η νομοθεσία πηγαίνει πέρα από τα όρια, κύριε Πρόεδρε. ουσιαστικά ε, με αυτή την ε, νομοθεσία ε, με τη Σέγγεν είναι απελευθερωμένη και η εμπορία ανθρώπων. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούν να παρέμβουν παρόλο που βλέπουν τι συμβαίνει διότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ατζέντα δεν επιτρέπει ε, τη χρήση συγκεκριμένων πραγμάτων. Όπως για παράδειγμα οι Ολλανδοί αστυνομικοί δεν μπορούν να παρέμβουν στα σύνορα γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ε εικόνες από βίντεο. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι ίδιοι οι άνθρωποι να παρέμβουν. Ελεύθερη κυκλοφορία, πολύ ωραίο πράγμα, αλλά είμαστε και λίγο αφελείς. Οι εγκληματίες όμως δεν είναι αφελές και, αφελείς και χρησιμοποιούν πλήρως οποιοδήποτε κενό προσφέρει νομοθεσία. Καλή και ωραία η Σέγγεν, αλλά αν έχουμε ορθά ανοιχτά σύνορα και δεν ελέγχει κανένα τα πράγματα, δεν μπορούμε να έχουμε λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φοντάνα για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για τη συμφωνία Σέγγεν, διότι πραγματικά βρισκόμαστε με ενώπιον μιας δύσκολης κατάστασης στις χώρες μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τους ελέγχους ε, στα σύνορα όταν υπάρχουν ε, ύποπτες μεταναστευτικές ροές. Μου φαίνεται και αυτή η κατεπίγουσα κατάσταση. Και σίγουρα είναι μια κατάσταση που ορισμένες φορές πραγματοποιήθηκε κιόλας διάβασα ότι σε περίπτωση κατεπίγουσας ανάγκης θα μπορούσαμε να έχουμε και ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα καθορίσει αν θα κάνουμε ελέγχους για δύο μήνες, για έξι μήνες και αν το πρόβλημα συνεχιστεί τι θα γίνει, θα σταματήσουμε και η οδηγία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται για χώρες οι οποίες είναι από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς ε, ε, εύρωστες. Κάποιοι πηγαίνουν σε άλλη χώρα για να εκμεταλλευτούν το κοινωνικό κρέτος. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν αποτελείται μόνο από καλούς πολίτες, ε, αποτελείται και από ανθρώπους που ίσως δεν έχουν και τόσο καλές προθέσεις. Και την εγκληματικότητα τι θα την κάνουμε. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι στα σύνορα. Σκεφτείτε ότι στη χώρα μου, για παράδειγμα, στην περιοχή του Βένετο, έγινε μία απόπειρα να επαναπατριστούν κάποιοι ε, κοινοτικοί υπήκοοι διότι ήταν κλιματίες, αλλά μετά από λίγο καιρό ε, ε, επέστρεφαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και ένα αντιστάθμισμα. Θα πρέπει να μπορούν να γίνουν επιστροφές και να μπορούν να γίνουν αποτελεσματικοί έλεγχοι στα σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ για δύο λεπτά εξ ονόματος της ε, Νοτικής Αριστεράς. Äh, Κυρίες και κύριοι, η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Είναι μία από τις ε, μεγαλύτερες και σημαντικότερες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν να αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Συνδέονται και με ένα άλλο θεομελαιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελεύθερη μετακίνηση. Διαπιστώνονται λοιπόν σημαντικές ελλείψεις. Ε, αυτό πρέπει να το πούμε. Και υπάρχει μια ειδική ρήτρα εσχάτης ανάγκης ε, αυτή αφορά στην αναχέτηση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι μετανάστες ε, είναι απλά η πρόφαση για να επαναφερθούν ε, οι συνοριακοί έλεγχοι, για να αιτιολογούνται Κατόπιν τούτου οι μετανάστες γίνονται οι αποδιοπομπέοι τράγοι της ευρωπαϊκής πολιτικής και αυτό είναι απαράδεκτο. Μετά από σύσταση του Συμβουλίου ε, μπορεί η ε, αναστολή, μάλλον η επαναφορά των ελέγχων να κρατήσει μέχρι και δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ο επόπτης ε, και το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε καν να εξασφαλίσει μια θέση στο τραπέζι σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν, εάν αυτή η πρόταση και το λέω αυτό ε, παρότι θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, δύο συγητές. Σας λέω λοιπόν ότι πράγματι για δύο χρόνια αγωνιστήκατε, αυτό είναι σωστό και χαίρομαι πάρα πολύ που προέκυψε τουλάχιστον ένας ε, μηχανισμός αξιολόγησης που φέρνει τη δικαιοσύνη ανάμεσα στα κρατημέλη και φέρνει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Παρόλα αυτά όμως έχουμε χάσει και ελπίζω αυτό να μην γίνει προηγούμενο για την ε, εκμετάλλευση του Κοινοβουλίου, των δικαιωμάτων μας. Ε, το Σέγκεν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις κατόπιν του για μας αυτό που έχει παρουσιαστεί δεν αποτελεί συμβιβασμό. Και τώρα μιλάμε πρώτος ο κύριος Ζήλστρα από το γραμμένο γραμμένος. Ε, βλέπουμε πως ε, τελικά το Σέγγεν ωφελεί περισσότερο τους ε, εγκληματίες και τώρα οι Βρυξέλλες πάλι γίνονται πιο ισχυρές και τα κράτη-μέλη πιο αδύναμα ενώ θα έπρεπε να επανεισαχθούν οι συνοριακοί έλεγχοι όταν το θεωρούν απαραίτητο τα κράτη-μέλη. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι ευχαρίστω δείχνουν το διαβατήριό του και εξάλλου ο έλεγχο του διαβατηρίου δεν θέτει σε αμφισβήτηση την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Γιατί λοιπόν είναι κατά όλη τη επανεισαγωγή των ελέγχων διαβατηρίων στα σύνορα. Το ΣΕΝΚ είναι μια πολιτική που έχει τελείω εκτροχιαστεί. Οπότε θα πω στα κατημέλη επιλέξτε το συμφέρον των πολιτών σας και ε, τελειώστε με αυτό το Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ομιλήτρια είναι η κυρία Ματιέ. Σας ευχαριστώ. Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Έχουμε κερδίσει διπλά. Καταρχήν, ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών ε, διατηρείται και είναι μια ε, θεμελιώδης ελευθερία γιατί δένει τους ευρωπαϊκούς λαούς και δείχνει μια απτή πτυχή της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Ε, γι' αυτό συζητάτε ως καλύτερη, μεγαλύτερη επιτυχία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Κάθε επαναφορά εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να γίνεται εκτάκτος μόνο σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου. Αυτοί οι έλεγχοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν μόνο την ε, ασφάλεια του χώρου Σέγγεν και άρα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε εξάλλου και έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πλέον αξιολόγηση ε, να βελτιώσουμε αντικειμενικά δε τους ελέγχους στα εξωτερικά μα σύνορα χάρη σε ε, επιτόπιε επισκέψει. Επίση, δώσαμε τα μέσα για να αντιδράσει κανεί τα εξωτερικά σύνορα και να ενισχύσει τους ελέγχου εκεί, ώστε ο πολίτη να μην αισθάνεται πω είναι διάτρητα αυτά τα σύνορα κράτη-μέλη θα μπορούν να αντιδράσουν και να ενισχύσουν τους ελέγχους σε, σε, σε, εφόσον διαπιστώθουν ελλείψεις. Θα είναι δε δυνατό η προσωρινή επανεισαγωγή ελέγχων σε εσωτερικά σύνορα για να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από ανεξέλεγκτες ροές. Όμως ιδιαίτερες ε, ε, περιστάσεις ε, μόνο όταν ισχύουν θα γίνεται αυτό. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επανεισάγουν εσωτερικούς ελέγχους για ε, λόγους ασφάλειας γιατί το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να προηγείται όλων. Είμαι πεπισμένη πως η διακυβέρνηση του Σέγγιν είναι μεγάλο βήμα μπροστά. Μα δίνει δε τον απαραίτητο μηχανισμό για να ελέγξουμε καλύτερα τα σύνορά μα. και χάρη σε αυτό θα εγγυηθούμε στου Ευρωπαίου πολίτε ένα χώρο Σέγγιν όπου θα μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν και αυτό με κάθε ασφάλεια. Αυτό το πακέτο το κερδίσαμε μετά από πολλέ μάχε και χάρη στο πείσμα των εισηγητών μα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ το Συμβούλιο σε αυτέ τι δεν είχε είχε πολύ δημοκρατική στάση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ματιέ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Γκέμπελς. Κύριε Πρόεδρε, το 1900 85 ήμουν από τους πρώτους που ζητούσα να υπάρξει η Συμφωνία Σέγγεν, μια συμφωνία την οποία δέχονται φυσικά και οι Ευρωπαίοι πολίτες και αγαπούν ιδιαιτέρως. Αρκετές ε, χώρες βέβαια ζητούν ρήτρε ε, διαφύλαξης ε, υποτίθεται με σκοπό να αντιμετωπίσουν τη λαθρομετανάστευση δεν θα πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή τη λογική, στο φόβο και στα εξωτερικά σύνορα και να χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα ότι ε, στα Ιταλικά, ε, στις Ιταλικές αχτές ε, καταφτάνουν πολλοί μετανάστες η συνθήκη Σέγγεν ήταν σαφής. Απουσία ελέγχων ανεξάρτητα από την ε, ε, εθνικότητά των Ευρωπαίων πολιτών όταν διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν τις συνθήκες. Υπάρχει κανόνας του 2003 ο οποίος επιβάλλει ότι σε κατεπίγουσα περίπτωση η οποία χαρακτηρίζεται ε, ως πολύ επικίνδυνοι, ο 118α, θα μπορούσαν ίσως να εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα επαναφοράς των ελέγχων. Αυτό και μόνο αρκεί και με το παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικές συνθήκες. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιες χώρες μέσω της συμφωνίας που ε, ε, συζητούμε τώρα είναι επανεθνικοποίηση των συνόρων και ε, είναι εκτός της παρούσας νομοθετικής διαδικασίας. Βεβαίως και η διαδικασία και η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ε, δίνει αρκετά σημαντικά στοιχεία. Λέει ότι αυτές οι διατάξεις θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσουν οποιαδήποτε ε, κίνηση είναι κατά των μεταναστών. Αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώνονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, μας δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως θα έπρεπε. Είναι εκατομμύρια οι πολίτε που διασχίζουν τα σύνορα. Ποιο μπορεί να του ελέγξει, Ποιο θέλει να σταματήσει του εκατομμύρια τουρίστες που θα επισκεφθούν φέτο το καλοκαίρι τη Γαλλία και την Ιταλία για παράδειγμα. Ποιο θέλει να σταματά κάθε μέρα του ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται σε γειτονική χώρα και διασχίζουν τα σύνορα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε όχι στη λογική του φόβου που έχει κυριεύσει κάποιε από τι κυβερνήσει μα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Σαρτζεντίνη. Because open here. I'm sorry. It is yeah. επιτέλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων επί συζητήσεων για το μηχανισμό αντίδρασης και τη δυνατότητα επαναφοράς ε, των συνόρων έστω και σε προσωρινό ε, επίπεδο μπορούμε πλέον να αποφασίσουμε. Ποιος κάνει τι όμως και πώς. Πλέον τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να πούν για ποιο λόγο θα ε, κλείνουν προσωρινά τα σύνορά τους. Δεν θέλουν να δεχτούν κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχουν στη συζήτηση. Κατ' εμέ, ο βασικός στόχος είναι να μπορούν να πούν στους πολίτες ορίστε, έχουμε και πάλι τον έλεγχο των συνόρων μας. Η Ολλανδική κυβέρνηση μια-δυο ώρες το μήνα ελέγχει τα δεδομένα ε, πολιτών ε, με ε, πινακίδες αυτοκινήτων της Ανατολικής Ευρώπης. Και αυτοί οι άνθρωποι αναφέρονται στο θέμα αυτό, λες και πρόκειται για ανθρώπους που υποκινούν την εγκληματικότητα και αυτοί οι άνθρωποι την χάνουν μεταχείριση σε εγκληματία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, ο κύριος Βλάσακ. κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Μιλάμε για το θέμα αυτό εδώ και πάνω από ένα χρόνο και η συμβιβαστική που επετεύχθη θα πρέπει να, να επιτρέπει μόνο σε περίπτωση απειλής της εσωτερικής ασφάλειας της εν λόγω χώρας την ε, επανεγκαθίδρυση ε, ελέγχων στα σύνορα και κυρίως μετά από συνεννόηση με τις ε, άλλες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου είναι ισορροπημένο αυτό το κείμενο και θα υπάρχει δυνατότητα να δούμε αν γίνονται μη εγκεκριμένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Οι Τσέχοι πολίτες έχουν αρνητικέ εμπειρίε, κυρίω όσον αφορά ε, τον έλεγχο από την γερμανική πλευρά των συνόρων. Θα πρέπει να υπάρχει νέο μέσο ε, για να ελέγχεται το σύστημα Σέγγεν χωρί ε, σύνορα στα εσωτερικά χωρίς ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μεγάλη επιτυχία και προ το κοινό μας συμφέρον θα πρέπει να κινηθούμε προς μια, ένα συντονισμό αποτελεσματικό με πλήρη ευθύνη όλων. Ο κύριος Μπάτεν για ένα λεπτό. Πέρσι είδαμε το σύστημα Σέγγεν να λυγίζει κάτω από την πίεση μαζικής μετανάστευσης και ορισμένα κράτη-μέλη επανεισήγαγαν μονομερείς ελέγχους. Η αναθεώρηση των κανόνων είναι ε, μια απόπειρα να κρατήσουμε το καπάκι πάνω σε ένα ντέτζερι που ζεματάει, αλλά είναι πολύ λίγη μικρή προσπάθεια και ανεπαρκής. Λέει ότι επιτρέπονται κάποια έλεγχη σε εξεκτακτές περιπτώσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πολύ λίγο και πολύ αργά. Ε, μία τέτοια πολιτική ανοιχτό σύνορο θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο μεταξύ χώρων με παρόμοια οικονομική και ε, πολιτιστική φύση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανοιχτά σύνορα είναι καταστροφική για τους απλούς ανθρώπους και έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Όλα αυτά έγιναν με την επιδίωξη μιας πολιτικής ιδεολογίας η οποία δεν είναι κοινή για τους λαούς της Ευρώπης και αυτή η ιδεολογία φυσικά είναι ότι η Ήπειρος της Ευρώπης είναι μία χώρα με Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, που δεν είναι φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτός τόπου και χρόνου και σε ένα πλαίσιο, ε, σε ένα διαγωνισμό ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην ιδεολογία, η πραγματικότητα πάντα κερδίζει. Ευχαριστούμε κύριε Μπάτεν. Κύριε Μπάτεν, ο κύριος, η κυρία... Είχατε μεγάλη επιτυχία. Δύο μπλε κάρτες προκαλέσατε. Μία από τον κύριο Γκέμπελς και η άλλη από την κυρία Μορβάη. τη δέχεστε? Ναι, βεβαίω, Γιατί όχι. Τέλεια. Κύριε Γκέμπελς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Μπάτεν μόλι είπε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ελέγχου των συνόρων είναι μια μεγάλη αποτυχία. Ξέρουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μέρος του χώρου Σέγγεν. Ο κύριος Μπάτεν μπορεί να μου εξηγήσει γιατί Υπάρχουν τόσο πολλοί λαθρομετανάστες στη Μεγάλη Βρετανία και γιατί η χώρα το που δεν είναι κομμάτι του Σέγγεν έχει τόσα προβλήματα με τους μετανάστες. Ωραία. Και τώρα η κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ πολύ. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Μπάτεν και τους υπόλοιπους δυτικοευρωπαίους φίλους μας, ως Ανατολικοευρωπαία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να επανεξετάσετε βασικά ολόκληρη την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και ανθρώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε, ε, σας παρακαλώ, να σκεφτείτε και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Οπότε, εμείς οι Ανατολικοευρωπαίοι ευχαρίστω να κλείσουμε ε, τα σύνορά μας μπροστά στο δυτικό κεφάλαιο και να πάρουμε πίσω την οικονομίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα έχετε κύριε Μπάτεν μου. Ναι, έλεγχη συνοριακή, λέει ο κύριο Γκέμπελ. Ναι, η Βρετανία είναι εκτό του συστήματο έγκαινα, αλλά υποφέρουμε από τι επιπτώσει του, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο να φτάσει στο καλέ και μετά να κάνει ένα άλμα στη Βρετανία. Και έχετε δίκιο ότι ακόμα και αν υποτίθεται ότι έχουμε συνοριακού ελέγχου εμεί, η μεταναστευτική μα πολιτική είναι αποτυχία στη χώρα μου και όχι μόνο λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω τη πλήρου ανικανότητα και τη έλλειψη βούληση τη Βρετανική κυβέρνηση να βάλει πραγματικού ελέγχου για του μετανάστε και να τους διεξάγει. Όντως αποτυχία στη χώρα μου που δεν οφείλεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας Μορβάη για την ελεύθερη κυκλοφορία των λαών, εμείς δεν πιστεύουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία των, την ελεύθερη κυκλοφορία των λαών στο κόμμα μου. Πιστεύουμε στην έλεγχο τη μετανάστευση και τη συνολική πολιτική. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε του μετανάστε ή να μην έρχεται πια κανένα, αλλά θέλουμε η δική μα κυβέρνηση να τα ελέγχει όλα αυτά προ το συμφέρον των Βρετανών, του Ιορδανικού λαού και όχι προς το συμφέρον μιας ιδεολογίας την οποία δεν συμμεριζόμαστε. Αν μπορεί κανείς να δεν ελέγξει τον κόσμο, είναι πολύ πιο εύκολο να το ελέγξει από ότι τα κεφάλαια που πολύ συχνά είναι μόνο νούμερα σε έναν υπολογιστή. Θα θέλαμε να υπάρξουν πολιτικές προς το συμφέρον του Βρετανικού λαού και μετά προς το συμφέρον των υπολείπων. Ευχαριστούμε κύριε Μπάτανα. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ομπερμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον ενθουσιασμό για το Σέγγεν. Ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει θετικέ ε, προτάσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα με όλες αυτές τις τρύπε που έχει στα σύνορα μοιάζει με ελβετικό τυρί το να θέλουμε να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας, καλό είναι αυτό, αλλά η απόφαση για την επαναφορά ελέγχων στα σύνορα, αυτό θα είναι θύμα της γραφειοκρατίας και το δικαίωμα για την επαναφορά των ελέγχων θα αφαιρεθεί από τα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι επίθεση εις βάρος της κυριαρχίας των κρατών μελών ε, για τη γραφειοκρατία. Υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τις όμορες χώρες ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν θα οδηγήσει πουθενά ή θα είναι πάρα πολύ αργά. Γιατί κυρίες και κύριοι οι λάτρομετανάστες δεν περιμένουν με υπομονή στα σύνορα μέχρι να αποφασίσουν οι Βρυξέλλες να δραστηριοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ούμπε Μάια. Και το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τελική συμφωνία για το πακέτο Σέγγεν συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο και την κυρία Βέμπερ για την προσπάθειά τους και να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι παρακολούθησα από κοντά και εγώ την όλη προσπάθεια ως εισηγητής για μια τρίτη έκθεση για την τροποποίηση και αναθεώρηση του κώδικα και, του, και της συνθήκης Σέγγεν σε άλλα σημεία, τα οποία ολοκληρώσαμε με τους συναδέλφους σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς κανένα πρόβλημα και την οποία ψηφίζουμε αύριο. Ο χώρος Σέγγεν και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου παραμένει μια από τις πλέον προωθημένες μορφές συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διέπεται από πολύ συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, πολύ δε περισσότερο απαιτεί το σεβασμό του από όλα τα κράτη μέλη. με δύο λόγια η ορθή διακυβέρνησή του η επιτυχία του εξαρτάται από την προσήλωση όλων των κρατών μελών και είναι προφανές πως μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τη συνολική προσπάθεια τραυματίζουν το αίσθημα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη που το απαρτίζουν συνολικά το χώρο σέγγεν. επομένω ανεύθυνε δηλώσει ή ακόμα και πολιτικέ διακηρύξει φανερώνουν απλώ άγνοια τη λειτουργία τη ευρωπαϊκή ένωση άγνοια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσων συμμετέχουν στι πιο προωθημένε ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα εκείνοι που για παράδειγμα πιστεύουν ότι δίνοντα ταξιδιωτικά έγγραφα σε παράνομου μετανάστε λύνουν το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών σε μια χώρα δεν γνωρίζουν αν έχουν αντίληψη τη πραγματικότητα, σίγουρα πάντω δεν έχουν καμία απολύτω γνώση και αντίληψη του πνεύματο και του τρόπου λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Δεν έχουν προφανώ καμία αντίληψη σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτών του στο λόγο. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα παρακαλώ, αν είναι εφικτό, να έχω μια απάντηση σε σχέση με το σημείο αυτό από την πλευρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βιώνει σήμερα την ε, ε, πρόοδο στο κοινό σύστημα ασύλου αλλά και στη δέσμη μέτρων για το Σέγγεν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για την λειτουργία των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγχαρώ λοιπόν τους εισηγητές οι οποίοι έφεραν σε αίσιο τέλος αυτά τα θέματα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να τονίσουμε τι ενίσχυση σημαίνει αυτό για τα κράτη-μέλη, για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ενισχύονται οι εξουσίες της ενημέρωσης ενημέρωσης και αξιολόγησης αυτής της τόσο σημαντικής δέσμης μέτρων για το κοινοτικό κεκτημένο και για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και κυρίως για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η δέσμη αυτή μέτρων ε, ε, προέκυψε μετά από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων λόγω των ε, λαϊκιστικών εκφράσεων που θέλουν την επανασυνικοποίηση μιας πολιτικής την οποία η συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά οριστικά και αμετάκλητα ευρωπαϊκή το μονομερές σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, ήταν ε, η συνέπεια αυτού του 1,5 χρόνου διαπραγματεύσεων που τελικώς καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε. Επομένως πρέπει να διαβεβάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιληφθεί του θέματος για οποιαδήποτε αλλαγή που θα προσπαθεί να γίνει στο μέλλον σε αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα. Θα διασφαλίσουμε την ε, ε, κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών και θεωρούμε ότι είναι από τους σημαντικότερους θησαυρού, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ευρωκοινοτικού κεκτημένου, διότι εκπροσωπεί την ελεύθερη κυκλοφορία 500 εκατομμυρίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό κυρία Κέλλερ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω αυτή η μεταρρύθμιση του Σάνκεν να συνεπάγεται πλονεκτήματα για του πολίτε. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι άλλο ένα λόγο γιατί να μπορούν να κλείνουν τα σύνορα. Υπάρχουν ελλείψει στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό μπορεί να σημαίνει τα πάντα, μπορεί και τίποτα. Επίση, και το ότι μια χώρα ενδεχομένως να δέχεται κάποιους μετανάστες μα αυτό είναι λόγος για να κλείνουν τα σύνορα με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι ελευθερίες στην Ευρώπη σε τελική ανάλυση η απόφαση είναι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών ε, παρότι ε, η απόφαση αφορά βεβαίως όλους τους Ευρωπαίους το Κοινοβούλιο στην αξιολόγηση δεν ε, παίρνει το ρόλο που το αξίζει θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την προσπάθειά τους αλλά σε τελική ανάλυση διαπιστώνω ότι δεν κατορθώσαμε να επιτύχουμε μια δημοκρατική αναθεώρηση του Σέγγεν και αυτό είναι κρίμα για τη τελική ανάλυση ο, το Schengen, ο χώρος του Σέγγεν είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αδιαμφισβήτητα, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει πραγματικά την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε άλλα κράτη-μέλη στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικές ε, οι προσωρινές ε, ανακλήσεις όταν υπάρχουν σημαντικές απειλές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές απειλές, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι ε, στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που αφορούν την ενίσχυση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για οικονομικούς λόγους. Εγώ θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές είναι αβάσιμες και δεν συνάδουν με τις κοινοτικές αρχές. Θεωρώ ότι δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, είναι ακατανόητες, ιδέως, ιδίως δεδομένων και των ωφελών που έχουμε για τους μετανάστες. Συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας που τους φιλοξενεί. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα, διότι υπάρχουν περιστατικά παράνομης μετανάστευσης και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπίλεν. Για ένα λεπτό ο κύριος Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αποτελεί σίγουρα κατάκτηση το σύστημα σέγγεν για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην ευρώπη. έχει όμως και παρενέργειες. είμαι από εκείνους που πιστεύουν στην αναγκαιότητα ασφάλειας των συνόρων των κρατών μελών που διασφαλίζεται βέβαια αποκλειστικά από την τήρηση και εφαρμογή των εσωτερικών κανόνων χωρίς παρέμβαση της ευρωπαϊκής ένωσης. υποτίθεται ότι επιχειρούμε να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη κατανομή του βάρους που ασκούν στις εθνικές κοινωνίες τα προσφυγικά ρεύματα. Πώς όμως εξασφαλίζεται αυτό κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι από τα 26 ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής Σέγγεν μόλις τα 6 δέχονται όλη τη μεταναστευτική πίεση ως χώρες των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βόρειες χώρες, οι χώρες που δεν έχουν θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που υφίσταται η Ελλάδα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό της. η οικονομία της χώρας μου και οι κοινωνικές δομές της έχουν κατακριουργηθεί και η ενεργεία έχει καλπάσει. δυστυχώς στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση δεν εμπεριέχεται καλόπιστος διαμοιρασμός ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη. αρκεί να σημειώσω το εξής ότι για την περίοδο 2007 χιλιάδες επτά έως σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μόνο στα έξι αυτά κράτη για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. το κόστος στην ελλάδα πάνω από 30 δισεκατομμύρια. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Όταν σας έδειξα το σφυράκι, βγάλατε δεύτερο χαρτί από ό,τι είδα. Την επόμενη φορά δεν θα σου το δείχνω το σφυράκι. Αστιεύομαι. Ο κύριος Γκόλνης είναι εδώ στην αίθουσα. Απουσιάζει. Ωραία. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κιγκαγκάλ. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμη συνάδελφοι, η συμφωνία την οποία πετύχαμε τις τελευταίες εβδομάδες περιλαμβάνει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα. Μπορέσαμε να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε το πιο σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεκτημένο δηλαδή Σέγγεν. Ελπίζουμε πως το καταστήσαμε πιο διαφανές και πιο αποτελεσματικό ταυτόχρονα και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κάρλος Κοέλιο και τον κύριο Βέμπερ για την εξαίρετή τους εργασία που δεν ήταν καθόλου απλή διαδικασία διαπραγμάτευσης και στο τέλος όμως όλα και τα τρία θεσμικά όργανα δέχτηκαν τα αποτελέσματα αυτά ως ένα βήμα μπροστά. Για να βελτιωθεί τώρα η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης ε, του Σέγγεν, που είναι ένας στόχος που πρέπει να υποστηριχτεί γιατί ενισχύει τα επιτεύγματα σε αυτό το τομέα για κάθε έναν από τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί υπάρχουν ε, ε, Υπάρχει δυνατότητα για την εισαγωγή, πανεισαγωγή μάλλον συνοριακών ελέγχων και η Κομισιόν μπορεί να είναι πιο δραστήρια όσον αφορά τις παρεμβάσεις της, αν στα εξωτερικά σύνορα ένα κρατος δεν είναι σε θέση να, ε, να επιτείνει τις προσπάθειές του. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη που είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκάλ. Μινούτο, la señora Guillaume. Η κυρία Γκυλιόμ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αλληλεγγύη και η αμοιβαία εμπιστοσύνη πραγματικά δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Η ελευθερία κυκλοφορία που πρόσφατα αφισβητήθηκε από διάφορα κρατημέλη, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να αποδείξουν, να αιτιολογήσουν τις, ε, ε, τους ισχυρισμούς τους για απάτη κοινωνικού τύπου. Ωστόσο, έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε με αυτό το συμβιβασμό στην ενίσχυση του κοινωνικού κεκτημένου και θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο Πρόεδρο, διατηρώντας ε, τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα θέμα που αγγίζει άμεσα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, τέλος, ε, να πάψει αυτή η αμοιβαία δυσπιστία και να ξαναβρούμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη που ίσχυε στην αρχή της δημιουργίας του Σέγγεν. Φαίνεται να όλα τα προβλήματα να, είναι, να οφείλονται τώρα στο κακώς διαχειριζόμενο γειτονικό κράτος και ελπίζω όλα αυτά πια να πάψουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιώμ. Για ένα λεπτό κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ. Η δυνατότητα ελέγχου των συνόρων είναι θεμελιώδης ε, για την εθνική κυριαρχία και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει ε, στην περιοχή του Σέγγεν. Εγώ συμφωνώ με την ε, πρόταση του Συμβουλίου ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να είναι των εθνικών κυβερνήσεων. Θα πρέπει όμως όλοι μας να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιες περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες μας και υπήρξαν και κάποια εκπληκτικά αποτελέσματα κάποιων ανθρώπων που μπόρεσαν να φύγουν από τη μία χώρα και διέπραξαν εγκληματικές πράξεις σε μία δεύτερη χώρα στην οποία ε, μετέβησαν και εκεί δεν ήταν και τόσο γνωστοί για τις πράξεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται πλήρης ανταλλαγή, ακριβής ανταλλαγή πληροφοριών. Η αντιμετώπιση των κινδύνων ε, που ε, ε, ε, μπορεί να προέλθει από ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνητικά επικίνδυνοι είναι πολύ σημαντική και ο έλεγχος των συνόρων μπορεί να βοηθήσει να επιτύχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μακοβέη τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω τις τρεις εκθέσεις του πακέτου Σέγγεν, διότι δημιουργούν ε, ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα οι βελτιώσεις που επιφέρουν αυτές οι εκθέσεις. καταρχήν προδιαγραφές για τα κράτη-μέλη Σέγγεν είναι πιο χαλαρές σε σχέση με τις υποψήφιες χώρες ε, όπως... Ε, ήταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά υπό το νέο σύστημα ε, οι κανόνε που θα ισχύουν θα είναι οι ίδιοι για όλου. είτε είναι υποψήφιε χώρε είτε ήδη μέλη τη Ένωση. Έτσι θα αυξηθούν οι προδιαγραφέ και θα υπάρξει και έλεγχο και εσωτερική έλεγχη, επιτόπι. Αυτή τη στιγμή Γίνονται παράνομα έλεγχοι διαβατηρίων στα εσωτερικά σύνορα πολλές φορές. Αυτό δεν θα είναι δυνατόν πλέον. θα μπορούμε να ελέγξουμε αν και ποιος μπορεί να εφαρμόσει ε, ελέγχους. Υπάρχει επίσης το θέμα της επανεισαγωγής συνοριακών ελέγχων σε ε, έκτακτες ε, περιστάσεις, αλλά μόνο μετά από συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν αιτήματος προς το Συμβούλιο Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας καλύτερος τρόπος προστασίας της δημόσιας τάξης. Ε, νομίζω πως όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ίδια για όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μωράες. Προέρχομαι, κύριε Πρόεδρε από ένα κράτος μέλος ε, το οποίο δεν ανήκει στο χώρο του Σέγγιν και αυτό προκάλεσε... Ε, εμείς λοιπόν έχουμε αναλύσει την πρόοδο που ανέφεραν οι δύο εισηγητές και βεβαίως ε, κατανοούμε και τις ε, αντιδράσεις στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίως όσον αφορά για το ότι δεν συμμετέχουμε στη συναπόφαση. Θέλουμε όμως να αξιολογήσουμε αυτά τα οποία πέτυχαν οι εισηγητές, το άλμα που έγινε από τον οπορτουνισμό και εγώ θέλω να κάνω την αξιολόγηση ως ένας πολίτης ε, ο οποίος ε, προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγμα το Σέγγεν το πρόοδο, διαφάνεια. Δεν είναι τέλεια η κατάσταση, όμως αποτελεί πραγματική πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου πολιτική ομάδα βλέπει θετικά αυτή τη συμφωνία. Πρόκειται για πρόοδο. Δεν είναι τέλεια η κατάσταση, αλλά εν πάση τόση είναι πρόοδος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μωράς. Κυρία Κολάσκα, Μπομπίνσκα. Ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, ήθελα να μιλήσω ε, μετά, αλλά κατά λάθο σήκωσα την πλέμου κάρτα. Για 1,5 λεπτό, κύριο Σκούρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τους συζητητές μας, τους συναδέλφους Κόγια και Βέμπερ, οι οποίοι εργάστηκαν ε, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία συζητούμε σήμερα. Καταρχάς ε, έχουμε τον μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης ε, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι διάφορε υπηρεσίε γίνονται πρωταγωνιστέ. Αλλά και για το γεγονό ότι συνειδητοποίησαμε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. Την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα έχω κατά νου σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε την αρχή τη ελευθερή κυκλοφορία, διότι είναι μία από τι βασικέ αρχέ τι οποίε στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και κάποια σημεία ε, τα οποία μα έδειξαν ότι υπάρχουν δυσκολίε. Υπήρξαν και δύσκολε στιγμέ στα κράτη κάτι μελη Δύσκολες όπως για παράδειγμα οι στιγμές οι οποίες προέκυψαν σε συνέπεια της ε, λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης. Και έπρεπε να παρέμβουμε και να ρυθμίσουμε τα πράγματα διότι υπάρχουν πολλές διαφορές στις κοινωνίες μας ήδη. Και όπου κάποιος ε, μπορεί να λάβει μονομερές αποφάσεις οι οποίες είναι ξαφνικές ε, μπορούν ε, σε κάποιες περιπτώσεις να διακυβεύσουν και την κοινή συμβίωση οι πολίτε μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών, χωρί αστυνομία, χωρί να χρειάζεται να επιδείξουν έγγραφα και αυτό ε, είναι η περηφάνεια μα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου. Και κάποιοι οι οποίοι ακούν αυτή τη συζήτηση από τα θεωρία να ρωτιούνται ίσως αν πραγματικά θέλουμε να επανέλθουμε σε ένα κόσμο ο οποίο δεν υπάρχει πια. Και εμεί φυσικά αυτό δεν το επιθυμούμε. Ευχαριστούμε κύριε Σκούρια. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μποσκούρτ. Δεν είναι εδώ η κυρία Μποσκούρτ. Ωραία. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Προτάσεβιτς. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η ελευθερία μετακίνησης χωρίς σύνορα, χωρίς διαβατήρια είναι μια από τις σημαντικότερες αποδείξεις για το ότι η Ευρώπη είναι πραγματικά ενωμένη. Αμφιβολία περί αυτού δεν υπάρχει. Ακόμη να γίνεται λόγος για δύο κανονισμούς. Ο ένας αφορά τις νέες διαδικασίες για την επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ελευθερία μετακίνησης. Και εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η κατεύθυνση των προτεινόμενων αλλαγών είναι ρηψοκίνδυνη. Δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο προτείνονται αυτές οι αλλαγές. Εγώ πάντως θα ψηφίσω υπέρ και των δύο εκθέσεων. Και αυτό θα το πράξω διότι πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά την επανεισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αλλά και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα δεδομένο κράτος πληρεί όλες τις απαιτήσει. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από κοινού και πρέπει να τα επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Και φαντάζομαι ότι και θα κοιτάζει πολύ προσεκτικά ε, Ω προ το κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι κανόνε ή όχι. Η μετανάστευση δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για την επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίε για πιθανές καταχρήσει. Διακόπτεται ο μιλητής. Ε, η κυρία Φλασίκοβα τώρα έχει το λόγο για μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή αφορά εγώ επανεισαγωγή ελέγχων στο Σέγγεν. Το 62% των πολιτών όμως της Ένωση θεωρούν ότι η ελευθερία κυκλοφορία μετακίνησης είναι μια επιτυχία και θα πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την ε, κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Πέρυσι παρατηρήθηκαν κάποια φαινόμενα. Και έτσι διακυβεύεται η ελεύθερη κινητικότητα. Κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει να φροντίσει να μην διακυβεύεται η ελεύθερη κινητικότητα. Η επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων υπό εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή. Θα πρέπει να αποτελεί μόνο μια ακραία λύση. Έτσι μια τέτοια απόφαση δεν επιτρέπεται να είναι απόφαση μόνο ε, ενό μεμονωμένου κράτου μέλου. Η αρμοδιότητα θα πρέπει να είναι τη ε, Κομισιόν και δεν θα πρέπει να αποκλείεται το Ευρωκοινοβούλιο από τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ως πολιτικός και ως ε, απλός πολίτης ε, θεωρώ το κεκτημένο Σέγγεν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό και να το εμβαθύνουμε περισσότερο. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις αρχές της ελεύθερης κινητικότητας. Εάν έχουμε τακτικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, αυτό θα αποτελέσει Όλοι θυμόμαστε πώς ήταν τα πράγματα τότε που πάντα υπήρχαν συνοριακοί ε, έλεγχοι. Αυτό επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί τώρα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η μετανάστευση είναι κάτι που υπάρχει, αλλά η αντίδραση σε αυτό δεν πρέπει να είναι ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα. Θα πρέπει να χειριστούμε με άλλο τρόπο το πρόβλημα. Η ελεύθερη κινητικότητα είναι μία από τις ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η κοινωνία μας. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, όχι να ε, ξαναεπιστρέψουμε στο παρελθόν. Και... Ε, έχουμε απομακρύνει πολλά ε, κράτη τα οποία θέλουν να, έχουν, ε, ε, να ενταχθούν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν εγγύηση της ασφάλειας, διαφάνεια και ευρωπαϊκό πνεύμα. Ο κύριος έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις δηλώσεις της ότι θα ήθελε να συμμετάσχει περισσότερο το Κοινοβούλιο και να τη συγχαρούμε καθώς και τους ομιλητές για το ρόλο, γιατί εξήρετο ρόλο της Ιρλανδικής Προεδρίας σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ε, δηλαδή το Σέγγεν και το ε, άσυλο. Και ελέγχ στην αρχή της Προεδρίας ότι η υπουργό θα παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε και αναφέρθηκε εδώ ότι το Συμβούλιο μια-δυο φορές ε, δεν παραβρέθηκε. Δεν παραβρέθηκε διότι δεν ε, κλήθηκε σε συμμετοχή. Υποστηρίζω τα μέτρα που προβλήθησαν. Θεωρώ ότι ότι το Σέγγεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ε, κίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, κεφαλαίων κλπ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι. Χρειάζονται ε, ασφαλείς έλεγχοι και μιλάμε και για μέτρα τελικής ίστατης καταφυγής, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέγιστο όριο πέντε ημερών καταρχήν και πιστεύω ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο που κινείται προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η αντίφαση από τις οποίες βρισκόμαστε τα επιχειρήματα και τα ενδιαφέροντα ε, όπως και συμφέροντα για το και είναι τεράστια και εντός και εκτός ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε συνέχεια η ουσία του να αντίθεται υπό αφισβήτηση που δεν είναι τίποτα άλλο από την απουσία εσωτερικών συνόρων εντός Ένωσης ε, και σε έναν ευρύτερο χώρο βέβαια. Ο λόγος ε, είναι μια ατέλεια, πολύ σημαντική ατέλεια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, πολύ απλή δεν εσωτερικεύσαμε, πολύ απλά σε επίπεδο κρατών μελών και αποτελεί, ούτε θα πρέπει να αποτελεί ένα νέο, έναν ενιαίο ε, χώρο. Γι' αυτό δεν δίνουμε και αρκετή στήριξη σε όσους ε, φιλούν ε, τα εξωτερικά μας σύνορα. Πηγαίνετε μια βολτά από τη Μάλτα από την Ελλάδα για να δείτε τι εννοώ. Και γι' αυτό προτιμούν να κλειδώσουν, να κλειδαμπαρωθούν τα κράτη-μέλη και όχι να εγγυηθούν την ελεύθερη διακίνηση σε όλη την Ένωση. Μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει δίκιο ε, που ε, τάχθηκε στα προτινόμενα, αλλά δεν είναι και αρκετά αυτά που προτείνουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος Γκεμπέλς και άλλοι. Ε, πόρο απέχουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς έχουμε τις καλύτερες δυνάμεις ασφαλείας και οι γείτονές μας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας που θα μπορούσε να απαιτήσει ένα κράτος μέλος. Ας σταματήσουμε και ας δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση ε, στο όλο αυτό ζήτημα, γιατί αλλιώς το Σέγγεν θα παραμείνει ένα πεδίο μαχών ε, μεταξύ των εθνικών κυριαρχιών. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Έγγελ. Για 1,5 τώρα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Παναγιώτοβα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Κοέλιο για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε με Κομισιόν και Συμβούλιο τη κανόνες διακυβέρνησης του Σέγγεν. Ε, σίγουρα ήταν ε, μακροχρόνιες και δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Στο μέλλον η αξιολόγηση ε, και ο σχετικός μηχανισμός για την παρακολούθηση του Σέγγεν θα είναι πιο πολύ ευρωπαϊκός. Καλό είναι να υπάρχουν τακτικές διαβουλεύσεις στις Κομισιόν με το Κοινοβούλιο ώστε να είναι πιο διαφανείς, απλοί οι κανόνες και το σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό. Εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί ο συντονισμό και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, γιατί ο χώρο Σέγγεν πάνω απ' όλα είναι ένα χώρο εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να δοθούν συλλογικέ λύσει, γιατί αυτέ είναι πάντοτε οι πιο αποτελεσματικέ. Νομίζω ότι έτσι θα αποτρέψουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ή κριτήρια σαν αυτά που εφαρμόζονται για την Ρουμανία και τη Βουλγαρία και θα βοηθηθούν οι δύο χώρε αυτές να προχωρήσουν στο Σέγγεν. Έτσι θα προωθήσουμε τη γεωπολιτική έννοια τη ασφάλειας στην περιοχή η Βουλγαρία. Τηρεί ήδη υψηλότατα πρότυπα συνοριακής ασφάλειας. Αν είμαστε μέλος του Σέγγεν θα αγγιηθούμε την ε, αξιοπιστία, την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ελπίζω η απόφαση για το Σέγγεν να μην αναβληθεί διότι αυτό θα θρέψει αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορεί η Ένωση τελικά να τηρεί τις δικές της αποφάσεις και δεσμεύσεις και ίσως ενθαρρύνει και ευρωσκεπτικιστικές τάσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Παναγιώτοβα. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και ο κύριος Ντίαθ Ντεμέρα έχει το λόγο ως πρώτος ομιλητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κάλλος και Ρενάτε. Σήμερα προχωρούμε ως προς την κοινοτική διάσταση του Σέγγεν μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας ε, διακίνησης των ε, πολιτών. Πρόκειται για μία ε, συνεχή και πολύ καλή εργασία και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Τα καταφέραμε πολύ καλά ως Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο ήταν άτεγκτο και άκαμπτο κατά τη διαδικασία. Θα έχουμε λοιπόν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την διαδικασία αποτίμησης και τη συνέχεια που θα δοθεί στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση η οποία σχετίζεται με τον χώρο ο οποίος απασχολεί τις αρμοδιότητες της κυρίας Μάλστρομ. Το Κοινοβούλιο πάντα θα υπαγρυπνεί και περιμένουμε πολύ περισσότερα από το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντίαθ Το λόγο έχει για ένα λεπτό Ευχαριστώ, λέει ο μιλητής. Είναι πολύ θετικό, θετικό το γεγονός ότι έχουμε μία ε, συνολική αντιμετώπιση του χώρου Σέγγεν, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Όμως δεν γίνεται τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λυθούν τα προβλήματα σε σχέση με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο χώρο του Σέγγεν. Τα ορισμένα κράτη-μέλη αντιτίθενται και αυτό αποτελεί κατάχρηση κάτι το οποίο μας απασχολεί μακροχρόνια. Η θέση αυτών των χωρών έδειξε ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, ανθίστανται παρά το γεγονός ότι υπάρχει κοινή ευθύνη. Και δυστυχώς μερικοί ευεργετούνται ενώ άλλοι όχι. Αυτές οι λαϊκιστικές τάσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αποδυναμώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι χάνουμε την αξιοπιστία μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή όλα τα κατάλληλα μέτρα ε, έτσι ώστε να, μπορέσει να, να μπορέσουν να διευρυνθούν τα σύνορα του Σέγγεν και να ε, μην υπάρχει αυτή η κατάχρηση. Ευχαριστούμε κύριε Λούαν. Το λόγο έχει ο κύριος Τζένκιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για... Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, για τη δουλειά που έχει γίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπερασπιστούμε μια πιο ε, ισχυρή ε, ζώνη Σέγγεν ε, και να υπερασπιστούμε και την Ευρώπη σε αυτές τις εποχές των ευρωσκεπτικιστών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη κινητικότητα και οι έλεγχοι στα σύνορα θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σήμερα είναι να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους στα ε, κράτη με εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι όχι μόνο τον συμφέρον των κρατών αυτών, αλλά είναι προ συμφέρον όλων των κρατών μελών. Και θα πρέπει γι' αυτό να βρούμε μία λύση ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί αυτοί οι έλεγχοι. Ευχαριστούμε κυρία Ζένκη. Κυρία Ζένκη, Η κυρία Ζασλοβιέκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή της Κομισιόν δείχνει με σαφή τρόπο ότι είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των ε, εξωτερικών συνόρων. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει πιο ευέλικτη η ζώνη Σέγγεν, ε, έχει να κάνει με το θεμελιώδες ε, δικαίωμα της ελεύθερης κινητικότητας και για λόγους εσωτερικής πολιτικής τα, κάποια κράτη-μέλη επιλέγουν να επανεισάγουν τους ε, συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Εάν ε, δεχτούμε όμως ε, αυτή την πρακτική, τότε ουσιαστικά θα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη βάση της. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τέτοιους ελέγχους και γι' αυτό στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να μπορεί η Κομισιόν να άρει τέτοιους ελέγχους. Θα πρέπει να υποβάλλεται ετήσια έκθεση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν. Και η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να πρόκειται για παρανόηση σχετικά με ε, τις ε, βίζες για τουριστικούς λόγους. Ε, οι τέτοιες πρακτικές δεν θα πρέπει να συνεχίζονται. Η παραβίαση της ζώνης Σέγγεν ε, με τουριστικές ε, θεωρήσεις ε, είναι κάτι το οποίο απειλεί την συνολική ζώνη Σέγγεν. Στην Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα φαίνεται ότι δεν αρκούν οι έλεγχοι που γίνονται και δεν ε, μας εκπλήσει και όλος ότι ε, τα νέα μέλη της ε, ζώνης Σέγγεν συχνά παραμελούν τους ελέγχους, δεν εφαρμόζουν επαρκώς και Γι' αυτό προσωρινή έλεγχη στα εσωτερικά σύνορα σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέλτσερ. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε που σήμερα αντί να συζητούμε για την προσχώρηση Βουλγαρίας-Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν, προσπαθούμε να αιτιολογήσουμε και να εξηγήσουμε και να συζητήσουμε για τους ελέγχους που λίγα, λίγα κράτη-μέλη θέλουν να πανησαγάγουν. Φαίνεται να κάνουμε δύο βήματα προς τα εμπρός και περισσότερα προς τα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους να πάψουμε το συντομότερο δυνατόν να μιλάμε για το κλείσιμο ε, για το άνοιγμα της χώρας Σέγγεν. Το Κοινοβούλιο έχει αποπροσανατολιστεί και έχει τεθεί και στο περιθώριο. Μέχρι στιγμής ο ρόλος του δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε. Δεδομένων των διευθετήσεων, πάλι θα συνεχίσει να είναι εκτός διαβουλεύσεων το Κοινοβούλιο, γι' αυτό θα στηρίξω την έκθεση, έχοντα βέβαια και μείζονες επιφυλάξει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, Εδώ κλείνει ο κατάλογο των ομιλητών με την κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εξαιρετικές περιστάσεις μπορούν να δικαιολογήσουν ε, αναστολή ενός από τα βασικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την ελεύθερη κινητικότητα των πολιτών. Σίγουρα το Κοινοβούλιο θα μπορεί να δεχτεί η επανεισαγωγή των ε, ε, ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπό εξαιρετικές περιπτώσεις, ε, εφόσον περιορίζεται η ελεύθερη κινητικότητα, εάν μπορεί να γίνει αυτό υπό εξαιρετικέ περιπτώσει, ε, γιατί ε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε και την ελεύθερη κινητικότητα των κεφαλαίων. Ε, εξαιρετικέ περιστάσει υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μου. οι μικρές επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ε, ανταγωνισμό απέναντι στο δυτικό κεφάλαιο. Ε, μπορούμε λοιπόν να περιορίσουμε και αυτή την κινητικότητα και να εισάγουμε προτιμησιακή μεταχείριση για τις επιχειρήσεις της χώρας λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων. Ευχαριστούμε. Κυρία Μορβάη, το λόγο έχει η Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν γιατί η Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν είναι θέμα συζήτηση σήμερα, αλλά θα επαναλάβω αυτά που είχε πει η Επιτροπή εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν τα τεχνικά κριτήρια και θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στο χώρο του Σέγγεν. Όμως ε, δεν είμαστε σε θέση εμείς να λάβουμε αυτή την απόφαση. Ελπίζω να ληφθεί στο εγγύς μέλλον. Η δημιουργία του Σέγγεν αποτελεί μεγάλο επιτεύγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 420 εκατομμύρια πρόσωπα κινούνται στα εσωτερικά σύνορα ε, με ε, τζίρο 1,5 δις ευρώ. Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να ταξιδέψει από τη, από τη Λετωνία, τη Φιλανδία μέχρι τη Μάλτα χωρίς να χρησιμοποιεί διαβατήριο είναι κάτι το πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα από τις διαπραγματεύσεις ότι θα θέλατε να έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα συμβασμό που ήταν ο μόνος εφικτός σήμερα και είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ελλείψεις στα εξωτερικά σύνορα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, διασφαλίσει ώστε τα κράτη-μέλη να μην προβαίνουν σε παράνομους ε, ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Γι' αυτό προωθήσαμε αυτή την πολιτική συζήτηση εδώ και 1,5 χρόνο. Θα πρέπει να μπορεί κανείς να ταξιδεύει εντός της Ευρώπης ε, χωρίς ελέγχους στα σύνορα σύνορα. Γι' αυτό θα ήθελα να υπερψηφίσετε τις ε, προτάσεις, τις δύο εκθέσεις, των Κουέλιο και Βέμπερ, που θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική εργασία τους, την οποία ολοκλήρωσα μέσα στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Κουέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την κυρία Μάλστρον. Στην ουσία από αυτή τη διαδικασία κερδίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εγκρίνουμε έναν κοινοτικό μηχανισμό. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες διορθώσεις σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν. Καταρχήν δεν ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει επανεισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό θα γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο με τη συνεργασία των κρατών μελών. Άρα δεν ελοχεύει κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν θα αποδυναμωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Ίσα ίσα θα ενισχυθεί γιατί εάν υπάρξει παράνομη εισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα τότε θα διώκονται από αυτό το μηχανισμό. Τρίτον, δεν ισχύει ότι η μετανάστευση οδηγεί στους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ε, απορρίπτουμε κάτι τέτοιο στο, στον, ε, με βάση το νομοθέτημα που θα εγκρίνουμε. Δεν πρόκειται για θέμα που αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστα μέρη του χώρου Σέγγεν. Αλλά δεν θα πρέπει πληρούνται οι Όρη, όχι μόνο τη στιγμή της προσχώρησης, αλλά και μετά τη στιγμή που θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αξιολόγησης, όλα τα κράτη-μέλη μόνιμα θα πληρούν αυτές τις συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αυτό το πρόσχημα κατά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, ακόμα και εκείνους που θα καταψηφίσουν, αλλά που μας ε, ενίσχυσαν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Έντσιου που μας ε, βοήθησε ιδιαίτερα και τη στενή συνεργασία με τη Ρενάτε Βέμπερ, την οποία ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Και η τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Βέμπερ, η δεύτερη συγκήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ε, χρησιμοποιήσω αυτά τα τελευταία λεπτά για να διαβιβάσω δύο μηνύματα. Καταρχήν, να ε, ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον φίλο και συνεργάτη, τον Κάρλος Κοέλιου και όλους τους σκιώδεις και συνεργάτες, καθώς και τους βοηθούς και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, σε μας, το οποίο μας βοήθησε ιδιαίτερα. Το δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να διαβιβάσω ε, είναι το εξής. Εγώ είμαι προευρωπαίστρια, όπως γνωρίζετε, και συνεπώς μία, από μία χώρα εκτός του χώρου Σέγγεν υπήρχε ε, στενή συνεργασία με μεγάλη αποφασιστικότητα γιατί θεωρώ ότι ο χώρος Σέγγεν ανήκει σε όλους τους Ευρωπαίους. Παράλληλα σκέφτηκα και τη χώρα την οποία εκπροσωπώ, τη Ρουμανία. Πιστεύω ότι αυτή η νέα διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν θα μας προλιάνει το το δρόμο για να μπορέσουμε να προσχωρήσουμε στο χώρο Σέγγεν, διότι το επιθυμούμε και θεωρώ ότι πληρούμε πλέον τους όρους. Θα θέλαμε κι εμείς λοιπόν να μπορούμε να έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βέμπερ. Κλείνει η συζήτηση επί αυτού του θέματος και θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30. Ε, Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο της μερικής μια κοινή συζήτηση για τις οικονομικές καταστάσεις και άλλα συναφή, ε, οικονομικές εκθέσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων με φόνη εκθέση Λένε και εκθέση Μακάρθη για τις περιποθέσεις διαφάνειας. Θα ξεκινήσω με τον εισηγητή κύριο Λένε, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 4 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε